Αγαπητοί συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση της Ολομέλειας. Καλώς ήλθατε. Χαιρετίζω και τον ε, κύριο Επίτροπο. Τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης έχουν διανεμηθεί όπως και τα κείμενα τα οποία έχουν εγκριθεί. Ε, υπάρχουν σχόλια για τα πρακτικά. Τα πρακτικά αυτά θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί.